Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση αλλάζει, βρίσκεται εν εξελίξη, κάθε ώρα έχουμε νέες πληροφορίες σε σχέση με αυτή την ε, διαφωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας βρίσκονται στα θεωρία. Τους καλωσορίζω ιδιαίτερα τον ε, κύριο Κεμάλ Αζίζ Σταμβουλέλ. Η Ινδονησιακή Αντιπροσωπεία φιλοξενείται επ' ευκαιρία της ε, συνεδρίασης της Διακοινοβουλευτικής ε, διάσκεψη Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδονησίας. Ξέρετε πώ πρόκειται για μια αναψώμενη οικονομία που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ΑΖΙΑΝ, την Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πρόκειται για την πρώτη χώρα με την οποία υπογράψαμε το 2009 Συμφωνία σύνδεση και Συνεργασίας και με μεγάλη ευχαρίστηση καλωσορίζω εδώ πέρα του Ινδονήσιου βουλευτέ. Επόμενο θέμα, προς ενημέρωση.